Μιλούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους. Λόγω πολέμων, φτώχειας, διαφθοράς, της ύπαρξης αυταρχικών ή απολυταρχικών καθεστώτων και ούτω καθεξής. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα έπρεπε να ενεργήσουμε στο επίπεδο ένωσης πιο έντονος, πιο, να γίνουμε πιο ορατοί και πιο συνεπείς ελπίζω, ώστε να ενισχύσουμε το σεβασμό των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις τρίτες χώρες. Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο πιο συγκεκριμένα, αυτό προσπαθώ να αναλύσω και να εξηγήσω στα πρώτα τρία κεντρικά τμήματα της έκθεσης. Το πρώτο τμήμα του κειμένου εστιάζει την προσοχή στα μέσα που χρησιμοποιεί η Ένωση για να προωθήσει τα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις τρίτες χώρες. Εξηγώ επίσης ότι οι ενέργειές μας μπορούν να έχουν περισσότερο αντίκτυπο εάν ε, καταφέρουμε να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητά τους, την αποδοτικότητά τους. Εδώ και κάποια χρόνια η Ένωση έχει αναπτύξει και ενισχύσει διάφορα μέσα τα οποία μπορούν να τις επιτρέψουν να επηρεάσει τις τρίτες χώρες για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας στρατηγικό πλαίσιο δράσης, ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα σημεία εστίασης που έχουμε φτιάξει στις αντιπροσωπίες μας. Πιστεύω πως η Ένωση έχει στη διαθεσή της μια ευρία πανοπουλία μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ήγηκε λοιπόν η ώρα η Ένωση να εστιάσει την προσοχή στην εφαρμογή όλων αυτών. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που ήθελα να διαβιβάσω στην πρώτη παράγραφο της ε, Εκθεση και όπως διαπιστώνετε αυτό το το πρώτο τμήμα υποδιαιρείται σε μικρότερα τμήματα γιατί είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για την ετήσια έκθεση που συντάσσουν η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, που υιοθετείται από το Συμβούλιο και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι πιο αναλυτική και λιγότερο περιγραφική. Χρειάζεται μια ανάλυση, όχι απλά μια περιγραφή, ένας κατάλογος δράσεων. Έπειτα προτείνω να εκφράσουμε τη γνώμη μας για το νέο πρόγραμμα δράσης που είναι ένα βήμα μπροστά αλλά που απαιτεί μεγάλη προσοχή και προσπάθεια ώστε η εφαρμογή του να είναι επιτυχής. Επίσης έχω αναθεωρήσει όλα τα μέσα, έχω εξετάσει μάλλον όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί η Ένωση για να προωθήσει τη δημοκρατία στον κόσμο το εντολή του ειδικού επισταλμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε χώρα, στα σημεία ε, επικέντρωση τη κατευθύνε γραμμή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτε καθεξή. Και εκεί έχω βάλει και συστάσει για κάθε ένα από τα σημεία. Πιστεύω πω πρέπει να κάνουμε συστάσει, τα οποία εν μέρει εντάσσονται, οι οποίε μάλλον εν μέρει εντάσσονται στι προτάσει που έχει συντάξει το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Θεωρούμε πως εν τέλει αυτό το κείμενο μπορεί να θεωρηθεί ως, ως ε, μέσο ε, προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και οι ε, επαφέ μέσω πολυμερών οργανώσεων και γι' αυτό και εστιάζει την προσοχή στο τέλος. Το μήνυμά μου είναι σαφές ελπίζω ότι δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατά το μέγιστο βαθμό πολιτικές που έχουν εξωτερική διάσταση για να ενισχύσουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία στι τρίτε χώρε. Αναφέρομαι βεβαίως στην εμπορική πολιτική και στην αναπτυξιακή πολιτική, αλλά και στην πολιτική διεύρυνση και γυρνίασης που πραγματικά περιέχουν ένα μεγάλο δυναμικό ώστε να συμβάλλουν με ποιοτικό τρόπο στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών. Όσον αφορά τώρα τη συμμετοχή μα σε πολυμερεί οργανισμού, η Ένωση και πρέπει να είναι δραστήρια, να είναι προσιλωμένη και τα κράτη-μέλη να ορίσουν μια κοινή ε, θέση όσο γίνεται πιο ε, γρήγορα, ώστε να υπάρξει αρκετό χρόνος για παρασκευαστικές συζητήσεις με τις τρίτες χώρες. Τα δύο άλλα τμήματα του σχεδίου έκθεση εστιάζουν στι δύο διαστάσει που αναφέρονται στον ίδιο τον τίτλο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και θέλω να τονίσω όλος ιδιαίτερο το θέμα της δημοκρατίας. Για το δεύτερο τμήμα, το κεντρικό τμήμα της έκθεσης, θα ήθελα να, επιμείνω σε κάποιους άξονες δράσης, επί των οποίων θα πρέπει να συνεχίσει να επιμένει η Ένωση. Η θανατική ποινή, η ελευθερία συνείδησης, η ανεξιθρησκεία, τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών είναι κάποιοι βασικοί άξονες που αναφέρονται στο πλαίσιο αυτό αλλά δεν θέλησα σε αυτό το τμήμα του κειμένου να αναφέρω όλα τα είδη των δικαιωμάτων που υπάρχουν και που είναι αναγνωρισμένα, ούτε να αναφέρω εξαντλητικά όλες τους άξονες δράσεις που πρέπει να ακολουθήσει η Ένωση. Όπως ανέφερα πριν από λίγο, στόχος μου δεν είναι να κάνω έναν ατέλειωτο κατάλογο και θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να μην προσπαθήσουν να, να πιέσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί στόχος της έκθεσης δεν είναι να έχουμε 100 σελίδες με καταλόγους και λίστες που τελικά θα είναι και ατελής. Αλλά να, έχουμε, να τονίσουμε κάποιου τομεί που θεωρούμε προτεραιότητα. Στο τελευταίο τμήμα δε, της έκθεσης ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας για το ότι η πρόθεση της δημοκρατίας μέχρι στιγμής έχει, έχει διατηρήσει δευτερεύουσα θέση στις πολιτικές της Ένωσης σε σχέση με τις ίδιες χώρες. Πιστεύω πως είναι σημαντικό η στήριξη της Ένωσης για τη διαδικασία εκδημοκρατισμού και παγίωσης της δημοκρατίας να είναι πιο σημαντική. Όπως λέμε και στην παράγραφο 75, η δημοκρατία με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αλληλένδετα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το ένα δίχως το άλλο. Αυτό είναι Η δημοκρατία θα έπρεπε λοιπόν ε, να, διατηρεί μια πιο σημαντική θέση και να σκεφτούμε αυτή τη δημοκρατία πέρα από την εκλογική διαδικασία βέβαια και βεβαίως και εκεί αυτή είναι πολύ σημαντική και το ξέρουμε όλοι αλλά θα πρέπει να περάσουμε πέρα από αυτό και να πούμε ότι το κράτος δικαίου, η δημοκρατία είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Η δημοκρατία, είναι εξαρτησία του δικαστικού σώματος, αλλά και η αμερόληπτη, αμερόληπτος δικητικός μηχανισμός και το καθεξής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ε, μιλήσουμε για εξωτερική μας ε, πολιτική προς τον ε, πληθυσμού, τους πληθυσμούς. Θέλουμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και τα δικαιώματα. Αυτά είναι τα θέματα που θα ήθελα να περιληφθούν στην έκθεση αυτή. Η βασική, λοιπόν μου ιδέα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει εφαρμογή και θα πρέπει να είμαστε και συνεπεί και ολοκληρώνω συνεπεί σε σχέση με του ίδιου μας εαυτού, όπως παραλέμε στην παράγραφο 3, ότι η εσωτερική και η εξωτερική συνοχή στην πολιτική της Ένωσης είναι σημαντική για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε σε διεθνές επίπεδο σε αυτά τα θέματα. Η συνοχή αυτή ιδιαίτερα δοκιμάζεται από την κρίση των προσφύγων που σοβεί, αλλά θα ήθελα να επιμείνω για το γεγονό ότι αυτή η έκθεση δεν είναι ο χώρο για να λυθεί αυτή η κρίση. Και θα ρίνω του αδέλφου να μην προσπαθήσουν να λύσουν την προσφυγική κρίση μέσω αυτή τη έκθεση. Η έκθεση αυτή δεν είναι η μία καλή ευκαιρία για να μιλήσουμε για τον σκοπό δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ίδια τα κράτη-μέλη. Αυτά αφορούν την ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Φυσικά και μας ενδιαφέρουν οι ανταλλαγές ε, απόψεων ανάμεσα στην Επιτροπή μας και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Αλλά να μην κάνουμε εμείς τη δουλειά τους. Ξέρω πως υπάρχει πάντοτε αυτός ο πειρασμός και θέλω να σας αποθαρρύνω ρητά γιατί σε αυτή την έκθεση πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην δράση της Ένωσης στις τρίτες χώρες. Αυτό είναι ο τίτλος και όλα της έκθεσης. Να κλείσω λέγοντας ότι με χαρά θα συνεργαστώ με τους κοιόδης εισηγητές που είναι σήμερα εδώ παρόντες. Η ανταλλαγή απόψεων έχει ήδη ξεκινήσει γιατί είχαμε επαφές με τους εκπροσώπους των κοινωνία των πολιτών αλλά και με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και θα σταματήσω με αυτά Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά θέλησα να συνοψίσω το περιεχόμενο και να αναφέρω το πλαίσιο αυτού του διαλόγου, έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε μια έκθεση ουσιαστική αλλά και ευανάγνωστη. Γιατί πιστεύω πως αυτό το χαρακτηριστικό είναι σημαντικό, δεν πρέπει να μετατραπεί η έκθεση αυτή σε μια μορφή που περιπλέκει τα πράγματα και μετά από ε, και να καταλήξουμε σε έναν αγώνα για να μπουν δύο-τρεις παράγραφοι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέδα. Τώρα, οι σκιώδεις εισηγητές. Δεν έχουμε χρόνο πολύ, όπως ξέρετε. Κυρία Πόστα από τους σοσιαλιστές πρώτα και μετά ο κύριος Δεσμάκερ από τους συντηρητικούς και μετά η κυρία Λόχμπιλερ από τους πράσινους. Σας παρακαλώ λοιπόν δύο λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, εκ μέρους του κύριου Παντσέρη που ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, θα σας μιλήσω τον αντικαθιστώ. Είναι σε αποστολή, κοινοβουλευτική αποστολή στο εξωτερικό. Μου έδωσε λοιπόν το σημείωμά του και θα σας το διαβάσω. Πρώτον λοιπόν, ευχαριστεί τον εισηγητή, τον κύριο Πρέντα, για το έργο του μέχρι σήμερα. Ως ε, τελευταίο εισηγητή το 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γνωρίζω πολύ καλά πόσο μεγάλη σημασία έχει η έκθεση αυτή και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλά και επικοδομητικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πάντα θεωρούσε την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για να αξιολογήσουμε όσο και για να ενημερώνουμε τους Ευρωπαίους πολίτες για την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επ' αυτού λοιπόν εκφράζω την ικανοποίησή μου που στο πρώτο αυτό σχέδιο υπάρχουν προτάσεις και ενδείξεις όσον αφορά κυρίως τον ρόλο των ευρωπαϊκών αντιπροσωπιών. Αναφέρεται και η ανάγκη κριτηρίων στις κατευθυντήριες γραμμές αναφέρεται ο έλεγχος και η αποτελεσματική εφαρμογή των ρήτρων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διεθνείς συμφωνίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες. Αναφέρεται επίσης η ανάγκη να προσέξουμε περισσότερο όσους αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πέρα από αυτά τα θετικά στοιχεία έχω και κάποιες παρατηρήσεις και όσον αφορά τη δομή και όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεση αυτή. Όσον αφορά τη δομή. Πρώτον, πιστεύω ότι η διάκριση σε κεφάλαια που κάνει ο συγγετής δεν είναι τόσο σαφής, είναι πολύ γενικά τα κεφάλαια και δεν υπάρχει σαφής διάκριση θεμάτων μεταξύ αυτών. Εγώ θα είχα προτιμήσει μια θεματική προσέγγιση όπως κάναμε και πέρυσι. Όσον αφορά το περιεχόμενο πρέπει να αναγνωρίσω ότι δεν αναφέρονται καθόλου ζητήματα που είναι προτεραιότητα τόσο για τους σοσιαλιστές όσο και στη διεθνή σκηνή για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Η ανατροφή γυναικών κοριτσιών, η σχέση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανάπτυξη, η σχέση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με διαφθορά, δικαιώματα των ΛΟΑΕΔΑ, αναπαραγωγικά δικαιώματα, δικαιώματα ατόμων με αναπηρία και δράση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα του κλίματος. Μια πρόταση ακόμα. Μπορούμε, αν θέλετε, το σημείωμα επίσης να το δώσουμε, ε? του κύριου Πενσέριου, οπότε ολοκληρώστε παρακαλώ. Ναι, ναι, βεβαίως. Οι περισσότερες τροπολογίε των σοσιαλιστών θα επικεντρωθούν σε αυτά ακριβώ τα ζητήματα. Είχαμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε και θα έχουμε και παρετέρω δυνατότητε να τα συζητήσουμε όλα αυτά στις συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Στενισμάκερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω μέσα στο χρόνο που μου δίνεται να πω τα σχόλια μου. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πρώτα απ' όλα για την προσέγγιση του. Την εκτιμώ ιδιαίτερα γιατί δεν πρόκειται για έναν ανοιχτό λόγο αλλά επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα ζητήματα και πιστεύω ότι είναι καλό αυτό. Θετικό. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή γιατί πράγματι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα κριτήριο για μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να παραμείνουν έτσι. Τα μέσα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο εισηγητής το είπε ότι η προσέγγιση είναι ακριβώς αυτή και εμείς αν πρέπει να υπογραμμίσουμε κάτι ε, θα σας πω ότι ήταν πολύ θετικό όπου αναφέρεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία ως μέσο που μπορεί να στηρίξει την κοινωνία των πολιτών στις γείτονε χώρες. Στην γραμμή λοιπόν αυτών που αναφέρατε κι εσείς, είμαι κι εγώ. Επίσης για έναν ευρύτερο μηχανισμό ο οποίος θα εποπτεύει τη δουλειά που γίνεται στα πλαίσια του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διάλογος ο οποίος πρέπει να αξιολογείται συνεχώς Επίσης, χρειαζόμαστε και πιο λειτουργικές κατευθυντήριες γραμμές. Έχουμε ήδη, αλλά πρέπει να γίνει κάτι πιο λειτουργικό. Συμφωνώ επίσης με τη θετική αξιολόγηση που γίνεται όσον αφορά τον ειδικό απασταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως υπάρχει και κάτι που με απασχολεί και με το οποίο δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και το ότι πρέπει να δούμε τη συνοχή ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική διάσταση. Μπορεί να μην είναι της παρούσης για την έκθεση αυτή, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Και το άκουσα και για το διάλογο που έχουμε και με την Λευκορωσία παίζει κάποιο ρόλο για την αξιοπιστία μας, για τη συνοχή. Διότι πολλές φορές κατηγορούμε χώρες εκτός συνόρων μας, αλλά ξεχνάμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνοχή εξωτερικό και εσωτερικό για να ενισχυθεί η αξιοπιστία μας. Ευχαριστούμε κύριε Ντεμεσμάκερ. Η κυρία Λόκβιλερ τώρα. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρεντά για την ε, τόσο πλήρη εκθεσή του. Και εκφράζω την ικανοποίησή μου επίσης και για την συνάντηση που οργανώνεσαι με την κοινωνία των πολιτών ο κύριος Πρεντά. Επί του περιεχομένου τώρα. Ιδιαίτερα όσον αφορά το χώρο της κοινωνίας των πολιτών και οι προθέσεις κάτω από τις οποίες δουλεύουν όσοι αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά είναι ζητήματα που πιστεύω ότι πρέπει να υπογραμμιστούν περισσότερο μέσα στην έκθεση θα υποβάλουμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Έπειτα, υπάρχουν και κάποιες θεματικές πολιτικές που αναφέρονται στην έκθεση μεν, αλλά η ομάδα μου θα ήθελε να επεκταθείτε περισσότερο. Όσον αφορά την μετανάστευση είναι ένα θέμα. Εδώ μπορούμε να δούμε και πράγματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τη διαχείριση συνόρων και το θέμα επίσης της μετεγκατάστασης. Κάτι άλλο είναι τα κοινωνικά δικαιώματα που πρέπει να έχουν πιο εξέχοντα ρόλο στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έπειτα το θέμα της ατιμορρησίας ή των ανθρωπιστικών ρυθμίσεων είναι πράγματα τα οποία αναφέρονται μεν στην έκθεση, αλλά θα ήθελα να επεκταθείτε περισσότερο. Και υπάρχουν και κάποια άλλα, τα οποία δεν αναφέρονται καθόλου στο σχέδιο. Εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν. Για παράδειγμα, ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία. Πρόσφατα εγκρίναμε μια πολύ καλή έκθεση πάνω σε αυτό το θέμα. Επίσης, το θέμα των Ιδρυμάτων των Εθνικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αντιτρομοκρατική πολιτική, το τράφικινγκ, η εμπορία ανθρώπων ελευθεροδιακίνηση, όλα αυτά είναι θέματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουμε σε διάφορες περιοχές και χώρες. Όπως επίσης τη σχέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την παραβίασή τους και τον αθλητισμό. Τέλος, το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Γιατί το σχέδιο αυτό έκθεσης ξεκίνησε το 2014 και θα εγκριθεί στα τέλη το 2015. Ίσως στο μέλλον πρέπει να καλύπτουμε τις ε, εξελίξεις στα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο μια συγκεκριμένη χρονιά, αλλά μέχρι τη στιγμή που θα εγκριθεί. Γιατί εδώ πρόκειται μόνο για το 2014. Νομίζω ότι θα ήταν πιο ενδιαφέρον κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε Λοκβίλερ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης ΑΦΚΟ. Ποιος εσείς ή... Θα δώσω το λόγο σε εσά πρώτα, επειδή δεν έχουμε αρκετό χρόνο, δεν σας πειράζει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον ε, εισηγητή για την ε, εξαίρεση εκθεσή του. εκθεσή του. Πολλά σημαντικά θέματα αναφέρονται εκεί. Αναγνωρίζω λοιπόν ότι έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο και αυτός και οι συνεργάτες του. Τώρα, πολύ σύντομα. Πρώτον, θέλω να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πρόγραμμα δράσης την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Όπως είπε και η κυρία Λοκπίλερ, Πρόκειται και το 2014 και είμαστε τώρα στο 2015. Ήθελα και εγώ να το πω αυτό. Δεύτερον, να διευκρινίσω λίγο την προσέγγιση μεσοδικαίου που αναφέρεται στην έκθεση. Είναι μια πολύ σημαντική αρχή βάσει της οποίας εργαζόμαστε. Πέρυσι εγκρίναμε μια εργαλειοθήκη, όπως την ονομάζουμε, για την προσέγγιση αυτή βασιδικαίου, με διάφορα μέτρα, διατάξεις τεχνικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο πρόγραμμά μας. Επίσης, θα δημιουργήσουμε και ένα πακέτο που θα συμπεριλαμβάνει την κατάρτιση των συναδέρφων βάσει αυτής της προσέγγισης ένα help desk από τις Βρυξέλλες για τους συναδέλφου που δουλεύουν επιτόπου στις διάφορες χώρες. Ε? Και θα τους προσφέρουμε επίσης και πράγματα γνωμοσύνη προκειμένου να μπορέσουν αυτήν ακριβώς τη διάσταση, μέσω δικαίου δηλαδή, να τη συμπεριλάβουν στο έργο τους. Ήτανε κάτι από τα πιο σημαντικά που κάναμε πέρυσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που όντως τώρα χρησιμοποιείται αλλά εξάντλησα και το χρόνο μου, οπότε θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Σικάρντο Σερή, επικεφαλής ε, του τμήματος ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς καλωσορίζουμε την έκθεση. Είχαμε καλές επαφές με τον κύριο Πρέντα τις τελευταίες εβδομάδες. Έχουμε προσωπικό που επεξεργάζεται την έκθεση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα λοιπόν για αυτή την ε, μορφή συνεργασία, τυπική μορφή συνεργασία και τον ενθαρρύνουμε συνεχίσει προς την κατεύθυνση αυτή όπως και να έχει. Εμεί είμαστε διευθυμένοι να συνεχίσουμε την υποστήριξη και το διάλογο που είχαμε μέχρι τώρα. Πολύ σύντομα μόνο. Για το περιεχόμενο συμφωνούμε με την προσέγγιση του κυρίου Πρέντα που καλύπτει πολλά θέματα χωρίς να είναι εξαντλητικός. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες συστάσεις, προτάσεις, ιδέες της ε, εκθέσεως και όσον αφορά τα δικά μας μέσα και νομοθετήματα. Ε, μέσα σε αυτή την ε, ισχνή, λιγνή θα έλεγα, μορφή νομίζω ότι προβάλλονται ακόμη περισσότερο από ό,τι θα συνέβαινε σε μια πιο εκτενή έκθεση, αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Ε, Λυθεύουμε ορισμένε από τι συστάσει αυτή τη στιγμή για την ετήσια έκθεση που δημοσιεύουμε κάθε χρόνο, βλέπουμε κάποιες συγκεκριμένε συστάσεις και όντως συμφωνούμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της ετήσιας έκθεσής μας, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε και βέβαια για το πρόγραμμα δράσης που όπως γνωρίζετε είναι το κύριο μέσο που έχουμε στη θέσή μας. Ξεκίνησε τον Ιούλιο και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης το προωθούμε. Βέβαια το κύριο θέμα τώρα θα είναι η υλοποίηση του ένα μέσων αρκετά εκτεταμένου. Επανέρχομαι λοιπόν για να πω ότι είναι αρκετές ενδιαφέρουσες ε, συστάσεις ε, για τα μέσα μας και θα, τα, τις συζητήσουμε σε επόμενες συνεδριάσεις για να προχωρήσουμε σε υλοποίηση τους προσεχείς μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν τόσο σύντομος και τόσο περιεκτικός και περιγραφικός. Ας περάσουμε λοιπόν στην ουσία την ε, γραμμή που επιλέγει ο κύριος ε, Πρέτα, την ακολουθούμε όλοι. Να είμαστε δηλαδή ε, ουσιαστικοί, συγκεκριμένοι, να εντοπίζουμε τα ζητήματα εγκαίρως. Πόσο χρόνο, 40 λεπτά κυρία Πρόεδρε, 40, 7 μάλλον, μάλλον προς το 7. Καλώς θα είμαι σύντομος και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της εξωτερικής δράσης, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, για τις τοποθετήσεις τους και της Επιτροπής βεβαίω για τις παρατηρήσεις όλες. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του αδέλφου Παντσέρη βεβαίως πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη υπάρχει περιθώριο βελτίωση της αφήνειας και είμαι από τους πρώτους που το πιστεύουν αυτό, διότι όπως έλεγα και πριν, πρέπει τελικά το αποτέλεσμα να είναι κατανοητό, ορατό. Γιατί αν κάνουμε κάτι το μη ορατό δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Α μην ε, παρασύρουμε σε ε, μία λάθος κατεύθυνση τους πολίτες, το κοινό μας, έτσι ώστε να μην τελικά διαβάζουν τίποτε, γιατί θέλουμε να έχουμε ένα κείμενο στεναρό ως προς το περιεχόμενο, ταυτόχρονα ευανάγνωστο, για να απευθύνομαι, απευθυνόμαστε και σε ένα ε, σύνηθες κοινό και όχι μόνο στον ειδικό. Και εκεί για να απαντήσω σε κάποιες τις ερωτήσεις της κυρίας Λόχπιλερ. Ασφαλώς θα προσθέσουν και οι συναδέλφοι από την Επιτροπή Ανάπτυξης κάποια πράγματα. Έχοντας αυτό υπόψη να απέφυγα να περιλάβω θέματα που φαντάζομαι θα εισαγάγει ο συνάδελφος Ντέβε. Ντέβα. Σχετικά με τα δικαιώματα και ζητήματα που έχουν εντοπιστεί από τους συναδέλφους της Επιτροπής Ανάπτυξης και καθώς είμαι και μέλος στην Επιτροπή Ανάπτυξη γνωρίζω ότι αναμένεται να καταθέσουν. Ευχαριστώ και τον κύριο Ντέμες Μάρκερ. Γνωρίζω πολύ καλά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία, European Fund for Democracy και ασφαλώς ε, στην αναζήτηση δημοκρατίας και αξιοπιστίας ε, είμαι και εγώ διαθέσιμος να ε, παλέψω για να βρούμε τα μέσα που θα μας το επιτρέψουν αυτό. Για την κυρία Λόχ την οποία επί τη ευκαιρία ευχαριστώ γιατί έδειξε ιδιαίτερη δραστηριοποίηση στο διάλογο που είχαμε με την κοινωνία των πολιτών. Μεγάλη χαρά συνεργάζομαι μαζί της. Θα πω ότι συμφωνώ λοιπόν ε, να συζητήσουμε κάποιες τροπολογίες που θα σήμαιναν καλύτερη εκπροσώπηση και παρουσίαση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και όλες τις άλλες, άλλες παρατηρήσεις. Καταπολέμηση της ατιμορρησίας, θεσμούς ε, διαχείρισης ανθρώπινων δικαιωμάτων, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και πολύ ευχαριστώ να συζητήσω μαζί σα όπως και με του άλλου συναδέλφου, λύσει που θα μα επιτρέπουν να μείνουμε σε αυτή τη φιλοσοφία, σε ένα κείμενο εύστοχο και ευανάγνωστο. Ευχαριστώ λοιπόν ε, τις υπηρεσίες όλες, οι Επιτροπής τη Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για την υποστήριξη και τις παρατηρήσεις τους, για την κυρία Λόχμπιλερ και την ερώτηση για το 2015. Εγώ φρόντισα να έχω ένα χρονοδιάγραμμα που θα μας επέτρεπε να ψηφίσουμε πριν το 2016, γιατί ε, εάν ψηφίσουμε το 2016 για μια έκθεση που αφορά το 2014 με τόσες εξελίξεις που έχουν παρισφρήσει, θα βρισκόμασταν σε δύσκολη θέση. Αυτό προσπάθησα να αποφύγω. Τώρα μπορούμε να επικεντρωθούμε ε, έτσι, για να βρούμε μια ισορροπία στο 2014 καταρχάς και να σημειώσουμε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη πρόσφατες εξελίξεις. Γιατί δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα τεκτενόμενα. Ίσως λοιπόν για το μέλλον βρεθεί μία λύση για να καλύψουμε πιο ξεκάθαρα και την περίοδο που καλύπτει η πρόταση για έκθεση επιτροπής και αντίστοιχα άλλα χρονικά ε, άλλες χρονικές μονάδες ή περιόδους ανάλογα με τις ανάγκες που θα επισημάνουν και οι λοιπές κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αυτά χαίρομαι βεβαίως για τις ε, συνομιλίες και τη συνεργασία με τους Σκιώδης και την περαιτέρω συνεργασία εδώ. Σας ευχαριστώ και στη συγγνώμη που μακρηγόρησα. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Τώρα έχουμε χρόνο για να περάσουμε στην ουσία των ζητημάτων. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία και όντως συμφωνώ να γίνει ψηφοφορία μέσα στο μήνα γιατί είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί το θέμα μέσα στο 2015, να ψηφιστεί μέσα στο 2015. Σας ευχαριστώ θερμά και τώρα πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Φάτου Μπενσούντα, εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου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 Thank Σας ευχαριστώ και καλώς ήρθατε σε αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με χαρά καλώς ορίζουμε την εισαγγελέα της Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κυρία Φάτου Μπενσούντα. Όλα αυτά χρόνια υπήρχε ο κύριος Μωρένο Κάμπο και άλλοι ανώτατοι Πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ποινικό δικαστήριο, η κυρία Μπενσούντα, εξελέγει από τη συνέλευση των ε, συμβαλωμένων κρατών τον Ιούνιο του 2012 μια συνενετική απόφαση. Ε, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ασχολείται με τα πιο περισσότερα διεθνή εγκλήματα, δυνάμει του άρθρου 5 του καταστατικού της Ρώμης, γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα ένοπλης επίθεσης. Το δικαστήριο έχει επανειλημμένως επιβεβαιώσει τη βούλησή του να επιβάλλει τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη και παρακολουθεί εκ του ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις δραστηριότητες του Διεθνούς Δικαστηρίου από τη στιγμή της σύλληψής του το Κοινοβούλιο ετοίμασε το 2011 μια κοινοβουλευτική έκθεση για να εκφράσει την υποστήριξή του στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψήφισμα το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η υποστήριξη προ το δικαστήριο με δράση πολιτική και διπλωματική. Η υιοθέτηση τη λόγω εκθέσεω ακολούθησε απόφαση της Επιτροπής, Υποεπιτροπής των Σπονών Δικαιωμάτων για την πρώτη εθνική διάσκεψη στη Ρώμη το 2010 στην Καμπάλα. Ε, το ψήφισμα για το έγκλημα επίθεσης του Ιουλίου 2014 συμπίπτει με την εκατοεντητηρίδα από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει, να υιοθετήσει μια κοινή θέση ε, για το καθεστώς της Ρώμης, για τη σύμβαση της Ρώμης και το Διεθνές Δικαστήριο και ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να, και τα κράτη-μέλη να υπογραμμίσουν την ε, οικουμενικότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου για την επιβολή της ποινική δικαιοσύνης ανά τον κόσμο. Και πριν δώσω το λόγο στην κυρία Μπενσούτα. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω μια αντιπροσωπεία εννέα μελών ε, βουλευτών για την παγκόσμια δράση, ένα δικτύου πάνω από 1.200 βουλευτών ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και πολλοί ευρωβουλευτές. Πρόκειται για ένα δίκτυο το οποίο ξεκίνησε μια εκστρατεία για την ε, κύρωση και υλοποίηση των, ε, του καταστατικού της Ρώμης για τη λειτουργία του Διεθνούς Δικαστηρίου. Καλώς ήρθατε και δίνω το λόγο στην κυρία Μπενσούντα. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου στην πρόεδρο της ε, Υποεπιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την κυρία Έλενα Βαρενσιάνο, την οποία εγώ αντικαθιστώ, λέει, κυρία Μπεσέρα. Θα ήθελε πολύ κυρία Παλεβέλενσιάρο να είναι εδώ, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι παρούσα. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να τη διαβιβάσετε την ευγνωμοσύνη μου για την πρόσκληση που μου απίθυνε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δραμάτισε ρόλο κλειδί για την ε, εξασφάλιση πολιτικής βούλης από τα μέσα της δεκαετίας του 90 σε υποστήριξη του, καθεστώ, του καταστατικού της Ρώμης και υποστήριξε το διεθνέ ε, Ποινικό Δικαστήριο από, την, ε, από το σχεδιασμό του ήδη. Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συμβαλόμενα μέρη στο καταστατικό της Ρώμης και θα ήθελα ιδιαίτερα να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για επικοδομητική συζήτηση θεμάτων κοινού ε, ενδιαφέροντος. Καθώς η Επιτροπή σας ασχολείται με μια ευρύτερη σειρά θεμάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προαγωγή του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αξιών σε τρίτες χώρες, και ενώ το πράγμα αυτό, θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτά τα θέματα πάνε χέρι με χέρι με ζητήματα που αφορούν την δική μου υπηρεσία, ιστορία των, ε, του Διεθνούς Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το καταστατικό της Ρώμης που θέσπισε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του 1948 είναι αλληλένδετη στενά. Ε, από τη δημιουργία λοιπόν του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έχει πάρει μεγάλη έμφαση ο όρος λογοδοσία και στο πλαίσιο των σοβαρών παραβιάσεων των δικαιωμάτων. Ε, το Δουπουδού, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ασχολείται με τα πιο σοβαρά εγκλήματα που αφορούν ε, τη διεθνή κοινότητα. Τα 123 συμβαλόμενα μέρη στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο έχουν δώσει την εντολή στην υπηρεσία μου για την διερεύνηση και την δίωξη των, ε, εις των ε, αυτούργων εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονίας και ενδεχομένω το δικαίωμα τη ένοπλης επίθεσης στο εγγύ μέλλον. Αυτή λοιπόν η δικαιοδοσία μπορεί να ασκηθεί ε, σε σχέση με εγκλήματα τα αποτρόπαια εγκλήματα που έχουν ασκηθεί στο ε, έδαφος των συμβαλωμένων κρατών ή από υπηκόου των συμβαλωμένων μερών, ανεξαρτήτως το που έχουν διαπραχθεί τα εγκλήματα, και μπορεί να επεκταθεί με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Εθνών ή με δήλωση από μη συμβαλόμενο μέρος που αποδέχεται την δικαιοδοσία του Δούπουδου. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε το Δούπουδου είναι προς το εθνικό ποινικό δικαιοδοτικό σύστημα και πάνω απ' όλα είναι ένα δικαστήριο ίστατης ε, καταφυγής ε, ή ένδικης προσφυγής. Το δικαστήριό μου μπορεί να παρεμβαίνει όταν τα συμβαλόμενα μέρη είτε ε, αρνούνται, είτε αδυναμούν να διερευνήσουν και να διώξουν εγκλήματα της αρμοδιότητας του Δουπουδού. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω μια ενημέρωση για το έργο της υπηρεσίας μου και για περαιτέρω, και προ, προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι βουλευτές του μπορούν να υποστηρίξουν την εντολή του της μου. Η υπηρεσία μου λοιπόν διεξάγει προκαταρκτικές προανακρίσεις σε, σε νέα περιπτώσεις Παλαιστίνη, Ουκρανία, Κολομβία, Γουινέα, Ιράκ για να σας δώσω μερικές ιδέες, προκειμένου να διερευνήσει αν υπάρχει ε, βάσιμο υλικό προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια ανάκριση. Αυτή η προανάκριση λοιπόν δεν αποτελεί ανάκριση, αλλά μόνο μια διαδικασία συλλογής στοιχείων που επιτρέπει στην υπηρεσία μου να προσδιορίσει ζητήματα ε, δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας και παραδεκτού. Ιδιαίτερα αυτό σημαίνει αξιολόγηση του τύπου και της βαρύτητας των καταγγελωμένων εγκλημάτων, εάν υπάρχουν γνήσιες ε, δικαστικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο κατά των ιδίων προσώπων, που θεωρούνται υπεύθυνα με βάση την δικαιοδοσία μας, και βέβαια με σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και της ε, σε εάν υπάρχει σε εθνικό επίπεδο ε, προχωρούμε εάν χρειάζεται τις έρευνες. Θα δώσω λοιπόν περισσότερε λεπτομέρειε. Έχουμε μια προανάκτηση για την κατάσταση στην Παλαιστίνη που συνεχίζεται ύστερα από την αποδοχή από πλευρά τη Παλαιστίνη, τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και τη προσχώρηση αυτή στο καταστατικό τη Ρώμη εφέτο. Το γραφείο μα λοιπόν, η εισαγγελία, προχωρεί με βάση την εντολή τη κάθε διερεύνηση με πλήρη ανεξαρτησία, αναλύοντα τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί από κάθε πλευρά, με πλήρη διαφάνεια και αμεροληψία, ε, ακολουθώντα τι. Ε, καθιστικές ε, πολιτικές και διαδικασίες. Η συνεχιζόμενη λοιπόν πρώτη φάση της προανάκρισης επικεντρώνεται στην συλλογή και ανάλυση πληροφοριών από κάθε αξιόπιστη πηγή. Για το σκοπό αυτό έχω εξ αρχής καλέσει κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να προσφέρει πληροφορίες και να συνεργαστεί με την εισαγγελία μας. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι έχει δοθεί ανταπόκριση στην έκκληση αυτή από όλες τις πλευρές της σύγκρουση και η υπηρεσία μας έχει μπορέσει να σημειώσει καλή πρόοδο. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό και είναι σημαντικό επίσης να συνεχίσει να προσφέρεται η ε, υποστήριξη στη δουλειά και στο, στην εντολή τη υπηρεσία μα. Σε σχέση με την Ουκρανία, λοιπόν, ξεκινήσαμε μια προανάξη τον Απρίλιο του 2014 επί τη βάση της πρώτης αποδοχής ε, της πρώτης δήλωσης αποδοχής από την Ουκρανία της ε, δικαιοδοσίας του Δουπουδού στις 21 Νοεμβρίου του 2013 έως τις 22 Φεβρουαρίου του 2014. Η πρώτη αυτή ανάλυση επικεντρώνεται στα λεγόμενα γεγονότα του Μαϊντάν, που έλαβαν χώρα κατά την ε, αυτή περίοδο. Όπω ασφαλώ θα γνωρίζετε, στι 8 Σεπτεμβρίου του 2015, πριν από μερικέ εβδομάδε, η κυβέρνηση τη Ουκρανία ε, προέβη σε μια δεύτερη δήλωση ε, ανάλογα με βάση το άρθρο 12 παράγραφος 3 του καταστατικού αποδεχόμενη για αυτή την περίοδο από 20 Φεβρουαρίου και ε, ε, εφεξής την δικαιοδοσία του Δουπουδού με βάση ή σε σχέση με καταγγελόμενα εγκλήματα διαπρεχθάντα επί της επικράτειάς της, χωρίς ημερομηνία λήξης. Επί τη βάση αυτή λοιπόν ξέτεινα το, προσωπικό, το προσωρινό χρονικό μάλλον πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης προανάκρισης για να συμπεριλάβω αδίποτε καταγγελόμενα εγκλήματα που θα μπορούσαν να έχουν διαπραχθεί στο ε, έδαφος της Ουκρανίας από τις 20 Φεβρουαρίου και εφ' τις 2014 και έφεξης, ε, με βάση την δήλωση αυτή. Δεν είναι λοιπόν συμβαλόμενο μέρος στο καταστατικό της Ρώμης Ουκρανία, αλλά με τελευταία αυτή δήλωση και χωρίς ε, ημερομηνία εκπνοής έχει αποδοχή την άσκηση της δικαιοδοσίας του Δουπουδού σε σχέση με εξελισσόμενα γεγονότα στην Ουκρανία. Υπήρξαν ε, εκκλήσεις από διάφορες πηγές για την, επικύρωση, για την κύρωση από την Ουκρανία του καταστατικού της Ρώμης που όσο άλλωστε αναφέρεται και στην Συμφωνία Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία. Από την ε, οπτική του δικαστηρίου θα ήταν ασφαλώς ε, πρόσδεκτη η εξέλιξη και ενθαρρύνω το Κοινοβούλιο να δει αν θα μπορούσε να συμβάλλει στην υποστήριξη της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση αυτή στην Κολομβία 24 Σεπτεμβρίου ο, η κυβέρνηση της Κολομβίας και η ΦΑΡΚ ε, προέβησαν σε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την περάτωση της συνεχιζόμενης ενόπλης σύραξης ε, που σοβεί εδώ και δεκαετίες στη χώρα. Η υπηρεσία μου καλωσορίζει κάθε ε, αντίστοιχη, ειλικρινή και πρακτική πρωτοβουλία που μπορεί να επιτύχει την ειρήνη, ε, θέτοντας τη δικαιοσύνη ως κρίσιμο πυλώνα μιας ε, βιώσιμης ειρήνης. Παρακολουθήσαμε λοιπόν ε, την ε, διαδικασία την δικαιοδοτική και τη δικαιοσύνη της Κολομβίας ε, και, την ειρήνη, και τις διαδικασίες ειρήνευσης εδώ και χρόνια και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να φτάσουν στη δημιουργία μιας ειδικής δικαιοδοσίας στα μέρη για την ειρήνη στην Κολομβία έχω σημειώσει με αισιοδοξία ότι η συμφωνία αποκλείει την χορήγηση ασδήποτε αμνηστίας για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και είναι σχεδιασμένη μεταξύ άλλων να θέσει τέρμα στην ατιμορρησία των πιο σοβαρών εγκλημάτων. Όταν ε, διατεθούν πλήρες πληροφορίες, η υπηρεσία μου θα τις ε, εξετάσει με μεγάλη προσοχή για να δει ε, τι θέση θα λάβουν στις συνεχιζόμενες προνακρίσεις μας. Για τις εξελίξεις αυτές, και ενώ βρίσκονται σε ένα πρώιμο στάδιο, είμαι πεπισμένη στην περίπτωση Κολομβίας, η λεγόμενη σκιά του δικαστηρίου, όπως κάποτε την απεκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, έδωσε ουσία σε αυτή την ευρέως αποδεκτή έννοια ότι η ατιμορρησία για ε, αποτρόπαια εγκλήματα και συλλήβδιν αμνηστεύσεις για τους υπευθύνους ε, δεν ισχύουν πια ως επιλογές. Στην περίπτωση Γουινέας είδαμε ότι η προκατακτική εξέταση, η προανάκριση δίνει την ευκαιρία για, στην υπηρεσία μου να συνεχίσει την ολοκλήρωση των στόχων της καταστατικού της Ρώμης και να ενθαρρύνει τις εθνικές διαδικασίες. Κατά την προανάκριση της 28 Σεπτεμβρίου 2009, για το, ε, της για, το, για τη σφαγή στο στάδιο Κόνακρη της 28 Σεπτεμβρίου του 2009, η υπηρεσία μας ιδιαίτερα έδωσε έμφαση και προσοχή σε πολυάριθμε καταγγελίες για εγκλήματα σεξουαλικού ή βασιζό, χαρακτήρα ή βασιζόμενα στο γένος, στο φύλλο και ιδιαίτερα ε, περιέγραψε μια σειρά από, παραγω, από παράγοντες όπως η υπηρεσία του ΙΠΑ του, του, του Ειδικού Εκπροσώπου των για τη σεξουαλική βία σε περίπτωση συγκρούσεων, σειράξεων και οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν συμβάλει στην ε, ενίσχυση αυτής της δυνατότητας των εθνικών αρχών. Έχουμε λοιπόν σημαντική πρόοδο, ε, απτή πρόοδο και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι απαραίτητη και ευπρόσδεκτη κάθε πρόοδος προς, το κράτος δικαίου. Η υπηρεσία μας παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάσταση στη Γουινέα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ ότι θα διστάσω να ανοίξω και ε, έρευνες ή ανακρίσεις για οποιαδήποτε από τις εννέα καταστάσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή σε προανάκριση, εάν κρίνω ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις του καταστατικού της Ρώμης. Η πλήρωση αυτών των κριτηρίων οδήγησε την υπηρεσία μου στην έναρξη ανακρίσεων σε εννέα περιπτώσεις. Ουγκάντα, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία σε δύο χωριστές περιπτώσεις, Σουδάν, Νταρφούρ, Λαϊκή Δημοκρατία του Καγκό, Κένια, Λιβύη, Ακτή του Ελεφαντοστού και Μαλή. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφέρω εδώ κάποιες από τις καταστάσεις αυτές που βρίσκονται σε ανάκριση ή έχουν ακόμη και προσαχθεί σε δίκη και ιδιαίτερα θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το δικαστήριο δεν είχε ποτέ το τόση δουλειά όσο έχει σήμερα. Ε. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι έχει πάρα πολύ δουλειά, όχι μόνο η δική μου υπηρεσία η εισαγγελία, αλλά επίση και η γραμματεία και οι δικαστέ. Η γραμματεία είναι αυτή η οποία προσφέρει τι κρίσιμε υπηρεσίε στου δικαστέ ε, και τα δικαστήρια, αλλά επίση και σε κάθε εμπλεκόμενο μέρο κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, καθώ και στου εκπροσώπου των θυμάτων. Στη διάρκεια αυτού του μήνα, λοιπόν, πολλά πράγματα έχουν συμβεί σε σχέση με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είχαμε τη δίκη τη ε, Μπόσκοντ Καγκάντα που ξεκίνησε στι 2 Σεπτεμβρίου, σημαντική δίκη μεταξύ άλλων, γιατί η εισαγγελία μα ε, πιέζει για την ερμηνεία του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου προκειμένου να, να συμπεριληφθούν και τα εγκλήματα σεξουαλικής βίας που διαπράττονται από ένοπλη ομάδα εις βάρος των μελών της. Με τη δίκη αυτή λοιπόν προσπαθούμε να κλείσουμε το χάσμα τιμωρησίας που είχε ε, δυστυχώς διαπραχθεί και που παραμένει ακόμη δυστυχώς σήμερα, έστω και αν είναι πιο αρές οι εκφάνσεις του πριν από δύο μέρες, 29 Σεπτεμβρίου. Άρχισε η δίκη σε σχέση με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κατά του Ζων Μπεμπά και άλλων. Αφορά ε, παραβιάσεις σε σχέση με την αποδοχή της δικαιοσύνης και ιδιαίτερα ε, παρενόχληση και καθυποταγή μαρτύρων. Τα, ε, πρόκειται για τις περίφημες 70 υποθέσεις, για τις περίφημες υποθέσεις του άρθρου 70 για τις υποθέσεις του άρθρου 70 ε, οι οποίες ε, μας επιτρέπουν ε, να παραπέμψουμε τους πέντε συγκατηγορούμενους και να αποστείλουμε ένα μήνυμα σε σχέση με τον σεβασμό της ανεξαρτησίας των μαρτύρων διότι έγινε απόπειρα για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Όσον αφορά τις συνεχιζόμενες ε, έρευνες, η πρόσφατη σύγκρουση της ε, Κεντρικής Αφρικανικής Δημοκρατίας, η υπηρεσία μου παρακολουθεί με ανησυχία τις βίαιες επιθέσεις που έγιναν τις τελευταίες μέρες ειρήνη είναι πολύ εθρευστή και ενώ συγκεντρώνεται η διεθνή κοινότητα στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να συζητήσει πώ θα σταθεροποιήσει και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτή τη χώρα, αυτά τα περιστατικά κινδυνεύουν να μα πάνε πολλά βήματα πίσω. Ο πρόεδρο Σάμπα Πάζα ηγείται μια σημαντική διαδικασία προ την ειρήνη και τη σταθερότητα, καθώ και τι δημοκρατικέ εκλογέ, βασίζοντα ε, την εργασία τη ε, κυρίω στον πυλώνα τη δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένου τη υποστήριξη για την εργασία του DPD. Θα ήθελα να συστήσω, να την ε, τιμήσω για το θάρρο και την αποφασιστικότητά τη και ελπίζω πω η Ένωση θα στηρίξει αυτέ τι προσπάθειε στην οικοδόμηση κράτου δικαίου στη χώρα που για τόσα πολύ ε, χρόνο υποφέρει από συγκρούσεις και τη βία. Στην περίπτωση του Μαλή, πριν από λίγες μέρες μόλις, ο Αχμάτ Αλμάχτη ε, παραδόθη στην ε, γίδα του δικαστηρίου από τις αρχές του Νίγηρα. Είναι η πρώτη περίπτωση στην έρευνα για το Μαλί και εστιάζει στην καταστροφή θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων. Το μήνυμά μας είναι σταθερό ότι πρόκειται για σοβαρά εγκλήματα και επίθεση κατά της ανθρωπότητας εν γέννη και δεν θα πρέπει να περάσουν ατιμωρητοί. Είμαι ευτυχής που η υπηρεσία μου μπόρεσε να συμβάλλει σε μια ενημέρωση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα τον Ιούλιο Πρόκειται όντως για ακόμα ένα ε, θέμα επί του οποίου η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συγκεντρωθεί ώστε να το αντιμετωπίσει και να το εμποδίσει. Να εμποδίσει τη διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων. Ε, οι βουλευτές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο προς αυτό, εξασφαλίζοντας ότι η νομοθεσία και οικονομική στήριξη θα υπάρχουν για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Αλλά θα ήθελα εν συντομία να τονίσω ότι στις 11 Νοεμβρίου στην ε, περίπτωση της εκτής του Ελεφαντοστού θα ξεκινήσει δίκη κατά του πρώην Προέδρου Λόρεν Μπάκμπο και του Τσάρλς Μπλε Ενώ η υπηρεσία μου πρόσφατα ξεκίνησε έρευνα και ανακρίσεις για τα εγκλήματα που διαπράχθησαν από την άλλη πλευρά της ε, σύραξης. Δυστυχώς αυτή η δεύτερη ανάκριση στην Κρήτη του Λεφαντιστού είχε καθυστερήσει για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως λόγω ε, λοιπόν πόρων και της ανάγκησε να γίνουν πιο αραιά οι διαθεστηριότητες οι ερευνητικέ τη υπηρεσία μου. Τέλο, στην Ουγγάντα η προετοιμασία για την επικύρωση τη καταγγελία και τη ακροαματική διαδικασία τον Ιανουάριο 2016 στην υπόθεση του διοικητή Ντομινί Κόνγκουεν του στρατού αντίστασης του κυρίου αυτό το προστίσαμε στην υπόθεση Μπέμπα, ε, που είναι η κύρια υπόθεση και περιμένουμε την απόφαση, καθώς και για την υπόθεση Κένια Ρούτο. Θα φαντάζεστε ότι θα συνεχίσω κατάπαυστα μέχρι ότου βρεθεί, ε, φτάσουμε στην ε, ε, λύση της υπόθεσης. Αυτή είναι μια πραγματικότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Δυστυχώς, ενώ υπάρχει γενικά στήριξη για το δικαστήριο, η αύξηση των υποθέσεων τελευταία χρόνια δεν ακολουθήθηκε από παρόμοια αύξηση πόρων. Ελπίζω πως η υποστήριξη που έδειξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν για τις δημοσιονομικές απαιτήσει του ΔΠΔ θα συνεχιστεί και για το μέλλον, μέσω δηλώσεων στήριξης ή μέσω συγκεκριμένων μέτρων μέσω της εθνικές ε, Δικαιοδοσίας και τους ε, υπεύθυνου για τη λήψη των αποφάσεων που ε, ευθύνονται για τον προϋπολογισμό. Δεδομένων όλων των υποθέσεων που πρέπει να ερευνηθούν και να διεκπεριωθούν οι υποθέσεις όλες αυτές, το ΔΠΘ μπορεί να είναι η πανάκια όσον αφορά την βία και τις σειράξεις. Τα κράτη θα πρέπει επίσης να φέρουν τις ευθύνες για την δίωξη των εγκλημάτων. Οι ευρωβουλευτές και, και οι βουλευτές εν γέννη φέρουν ευθύνη γιατί πρέπει να εξασφαλίσουν ε, τους απαραίτητους πολιτικούς και οικονομικούς πόρους ώστε να διεκπαιρεώνονται αυτές οι υποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη του κράτους δικαίου, εκεί όπου και διαπράττονται κλίματα τύπου του, για το οποίο είναι υπεύθυνο το ΔΠΔ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός εταίρος στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας. <coughs> μέσω της στήριξης στις τρίτες χώρες και της άμεσης στήριξης. Επ' αυτού λοιπόν, σημειώνω με ιδιαίτερη εκτίμηση την βοήθεια που μας δίνεται για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η στήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι ζωτική σημασία προκειμένου να υπάρξει συνδυτοποίηση του κόσμου και προκειμένου η διεθνής ποινική δικαιοσύνη να εγκαθιδρυθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έχουμε σημειώσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δυσαρέσκεια να διακόψει τις ε, χρηματοδοτικές ευκαιρίες για μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις που προμοθούν το ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο έχει σοβαρές συνέπειες και όσον αφορά την προβολή των θυμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και όσον αφορά το πολιτικό επίπεδο την πολιτική στήριξη δηλαδή που τόσο πολύ χρειάζεται το δικαστήριό μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές έχει εκφράσει την ανησυχία του για παραβιάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καταστάσεις που έχουν να κάνουν με θέματα που εξετάζει το δικαστήριο. Επίσης, καταλαβαίνουμε τα διάφορα ζητήματα που ατομικά επιμέρους κράτη-μέλη θέτουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Θέσης όσον αφορά τις ε, δραστηριότητες του στήριξης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Πάντως, Σίγουρα χρειάζεται συνειδητοποίηση όσον αφορά τις παραβιάσεις που γίνονται, όσον αφορά το θέμα της λογοδεσίας και όσον αφορά την προβολή θεμάτων διεθνούς δικαιοσύνης. Θέλω να θαρρύνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να μας στηρίζει, γιατί χρειαζόμαστε και, πολιτικό και, και πολιτική και διπλωματική στήριξη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ζωτική σημασία για την ε, υπηρεσία μου, για την εισαγγελία δηλαδή του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου και προκειμένου να μην υπάρχει ατιμορρησία. Εξαρτώμεθα από την συνεργασία μας με άλλες πλευρές. Για παράδειγμα, το δικαστήριο εξαρτάται από τις χώρες μέλη προκειμένου να ε, μπορεί να συλλαμβάνει ε, υπόπτους είναι ένα θέμα βέβαια πολύ ευαίσθητο το θέμα των φυγάδων, αλλά γι' αυτό ακριβώς και χρειαζόμαστε πολιτική στήριξη από τη διεθνή κοινότητα και και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί εταίρο κλειδί για πολλές χώρες. Εδώ πρέπει να πω ότι η Νότια Αφρική δεν βοήθησε προκειμένου να συλληφθεί ο Αλ Μπασίρ στην ε, διάσκεψη που έλαβε χώρα στο Johannesburg τον Ιούνιο. Δυστυχώς τα θύματα των εγκλημάτων που έλαβα χώρα στο Δαρβούρ θα πρέπει ακόμα να περιμένουν, γιατί οι υπεύθυνοι δεν θα πάνε γρήγορα στη δικαιοσύνη. Επίσης υπάρχει και υποχρέωση των χωρών να εφαρμόζουν τα δάλματα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και είναι κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί και από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αλλά και από το Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Ενώ λοιπόν η συνεργασία και η στήριξη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ Ήτανε κάτι μάλλον απογοητευτό. Τώρα βλέπουμε και εγώ και η υπηρεσία μου ότι χρειαζόμαστε στήριξη για να πετύχουμε τους στόχους μας με τις δικές σας δράσεις. Διότι θα πρέπει αμερόληπτα και με συνέπεια να στηρίζουμε τις αρχές μας δρούμε σε ένα διεθνές και περίπλοκο περιβάλλον με διαφορετικά συμφέροντα που διακυδεύονται. Και μερικές φορές οι πολιτικές και οικονομικές, τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα θα έλεγα πιο πολύ, έχουν συνέπειες. Γι' αυτό λοιπόν όπως ε, εμείς εφαρμόζουμε την ίδια νομοθεσία και τις ίδιες προγραφές σε όλες τις περιπτώσεις, όσοι στηρίζουν το δικαστήριό μας πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι δεν είναι δυνατόν να ζητάμε την παρέμβαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε μια περίπτωση όταν αυτό τους βολεύει και να το αρνούμεθα σε κάποια άλλη περίπτωση, γιατί έτσι διακυδεύεται η ίδια αξιοπιστία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Άρα λοιπόν σε μερικές περιπτώσεις ε, θέλετε την ε, δίωξη, σε άλλες όμως όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να φαίνεται σαν να μεροληπτεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και χάνει την νομιμότητά του. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, υπηρεσία μου είναι μια μεγάλη πρόκληση προκειμένου να πετύχουμε λογοδεσία και δικαιοσύνη υπέρ των θυμάτων των πιο αποτρόπιων εγκλημάτων που γίνονται σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει να βάλουμε μαζί τις προσπάθειές μας προκειμένου να στείλουμε ένα σημαντικό μήνυμα με συνέπεια όσον αφορά την ανθρωπότητα για την ατιμορρησία και για το ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρούνται. Αυτή είναι μια πρόκληση που καμία χώρα και κανένας οργανισμός δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και εκφράζω την ικανοποίησή μου όσον αφορά τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών του, των Ευρωβουλευτών δηλαδή, και σας ενθαρρύνω να βρείτε και άλλους τρόπους να στηρίξετε το έργο μας. Προσβλέπω σε συνεχή συνεργασία μεταξύ μας, μεταξύ όλων μας και ελπίζω ότι η υπηρεσία μου μπορεί να συνεχίσει να στηρίζεται στη δικιά σας υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πολύ εκτεταμένη και ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Θα δώσω το λόγο στον του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Δεμεσμάκερ, η κυρία Άουκεν, ο κύριος Καστάλντο. Και σας καλωσορίζω. Αν μπορέσετε να περιοριστείτε στα τρία λεπτά, θα είναι πολύ καλό. ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω, αλλά όπως καταλαβαίνετε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι τόσο σημαντικό όργανο. Θέλω να ευχαριστήσω την προσκεκαλυμένη μας για την επίσκεψή της εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ομάδα μας πρέπει να ξέρετε ότι στηρίζει απόλυτα την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το ε, Διεθνούς Ποινικό Δικαστήριο που είναι μοναδικό στη φύση του. Έχω όμω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα για την ε, Ουκρανία. Οι Ουκρανοί έχουν κουραστεί, βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση και θα ήθελαν οι υπεύθυνοι για τη σφαγή της Μαϊντάν να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν. Οπότε, τι δυνατότητες βλέπετε, εντάξει, εξαρτάται και από τη συνεργασία με τη Ρωσία προφανώς, αλλά εσείς πώς βλέπετε εδώ τα πράγματα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι μέλος αντιπροσωπείας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ουκρανία. Και εμείς πιέζουμε τους συναδέρφους στην Ουκρανία να επικυρώσουν την ε, Σύμβαση της Ρώμης. Πιστεύουμε ότι θα είναι θετικό. Έρχομαι τώρα στην Παλαιστίνη. Εδώ βέβαια είναι θέμα συζητήσιμο. Η Παλαιστίνη είναι μέρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ανακοίνωσαν αμέσως ότι τους εγκληματίες πολέμου στη Γάζα θα τους φέρουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά βέβαια οι Ισραηλινοί δεν το πήραν καλά. Για μας, εμείς στηρίζουμε το δικαίωμα της Παλαιστίνης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο γιατί για μας το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν μεροληπτεί υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Για μας διεθνώς αναγνωρίζεται γιατί καταπολεμά την ατιμορρησία. Η ειρηνευτική διαδικασία βέβαια είναι σημαντική συγχρόνως στην περίπτωση της Παλαιστίνης, οπότε ρωτάω. Βοηθάει την ειρήνη κάτι τέτοιο και την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ ή όχι κάτι τέτοιο. Άγιες και Συρία. Η Συρία δεν είναι μέρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά ο κόσμος αναμένει ότι οι εκεί εγκληματίες ε, πρέπει να διωχθούν και να τιμωρηθούν. Συνεπώς, τι δυνατότητες υπάρχουν γι' αυτό. Μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας αυτό. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Είδατε και την ε, στάση της Ρωσίας. Ή μέσω καταγγελίας όσων ε, συμμετέχουν στο ΑΙΕΣ, στο λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Μήπως έτσι μπορούν ε, να πάνε στο δικαστήριο, να καταγγελθούν. Και κάτι ακόμα για την Νότια Αφρική και το γεγονός ότι ο Σουδανός πρόεδρος ξέφυγε και μπήκε στο αεροπλάνο τη στιγμή ακριβώς που γινόταν η ακρόαση στη Νότια Αφρική. Τέτοιου είδους ε, καταστάσεις πώς μπορούμε να τις εποφύγουμε στο μέλλον. Μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε κάτι άλλο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ τον όλα. Υπάρχουν δηλαδή χώρε οι οποίε αποτελούν μέρο του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου που βοηθούν κάποιον να ξεφεύγει. Πώ πιστεύετε εσεί ότι πρέπει να λειτουργήσουμε ώστε να τα καταφέρουμε καλύτερα σε αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Δενισμάκερ. Η κυρία Όκεν. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κυρία Πρόεδρε. Χάρηκα που σας άκουσα. Θέλω τα σχόλιά σας παρακαλώ για το εξή. Για πρώτη φορά στην ιστορία η στήριξη του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους δεν ε, ακολούθησε δήλωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά που θέλει η Παλαιστίνη. Εσείς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει κάπως το θέμα αυτό της Παλαιστίνης το λεγόμενο Ισλαμικό κράτο. Θέλω τα σχόλιά σας από αυτού και έχω και μια ερώτηση για φέτος. Πώς βλέπετε εσείς την προκαταρτική εξέταση για την Παλαιστίνη, πόσοι υπάλληλοι δουλεύουν πάνω σε αυτή την υπόθεση και πώς αξιολογείται τη συνεργασία με το ΠΙΕ και τις Παλαιστινιακές Αρχές είναι σημαντικό εσείς να πάτε στην Παλαιστίνη πριν ολοκληρωθεί η προκατακτική εξέταση. Το Παλαιστινιακή Αρχή. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από τον είπα εκπρόσωπο να δουλέψει για την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων που έγιναν στην Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ όσον αφορά την σύγκρουση στη Γάζα του 2014. πώς εσείς θα προχωρήσετε στην περίπτωση που δεν υπάρχει συνεργασία από κάποια από τις πλευρές. Έπειτα, δεδομένου ότι είναι περίπλοκη η κατάσταση και τα πολλά εγκλήματα τα οποία έχουν λάβει χώρα, πού θα επικεντρωθείτε στην προκαταρτική εξέταση. Τέλος. αναμένετε κάποια εξωτερική πίεση κατά τη διάρκεια της προκαταρτικής σας εξέτασης. Και υποσχέθηκα στην Μπάρμπαρα Λόκκριτ να υποβάλω και τις δικές της δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, ευθυγραμμίζεται βέβαια με αυτά που είπα και εγώ, αλλά είναι και πιο γενική. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει παραπάνω η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σας στηρίξει. Και δεύτερον, έχετε τη συνεργασία που χρειάζεστε για να προσφέρετε δικαιοσύνη στα θύματα. Και θέλει επίσης να ξέρει, αλλά και εγώ, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις όπως είναι αυτή της Συρίας. Όπου θα μπορούσε ίσως να κάνει μια προσφυγή το ποινικό διεθνές δικαστήριο. Ευχαριστούμε κύριο Καστάλντο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ Θέλω να ευχαριστήσω και την εισαγγελέα Μπεν που βρίσκεται σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη τιμή για την Επιτροπή μας αλλά και για το Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ τη συνεργασία με το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Το είπατε προηγουμένω και το επαναλαμβάνω και εγώ. Μπορώ να σα διαβεβαιώσω από πλευρά μου αλλά και από πλευρά άλλων συναδέλφων αλλά και από ολόκληρο το Κοινοβούλιο, από τη δική μας πλευρά, η όθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο θα πιέσουμε ώστε να προωθηθεί το, κοινο, το δικαστήριο αλλά και να έχει τις πλήρες δυνατότητες ώστε να αποδώσει δικαιοσύνη. Για παράδειγμα στην Ιταλία το λέω με μεγάλη πικρία. Η χώρα μου ακόμα δεν έχει επικυρώσει τις τροπολογίες της Καμπάλα μαζί με έναν συνάδελφο ζητήσαμε γραπτός ε, νομοσχέδιο για να πιέσουμε την κυβέρνησή μας να κυρώσει τις τροπολογίες. Είμαστε λοιπόν ε, ε, σταθερά υπέρ. Όμως και άλλοι συναδελφοί θα, ανέφεραν και θα θέλαμε και εμείς να επέξετε πιο αποφασιστικό ρόλο όσον αφορά τα εγκλήματα που έχουν γίνει στην Παλαιστίνη. Δεν μιλάμε εδώ για κάποιο μηχανισμό Βεντέτας. Πρόκειται όμως για δύο λαούς που και οι δύο ζητάνε δικαιοσύνη. Το να μεταφερθεί αυτό το πλάνο από το διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο που φαίνεται να έχει μπει σε ένα φαύλο κύκλο σε έναν τέτοιο μηχανισμό, στα όσα προβλέπει το καθεστώς του δικαστηρίου, θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να, βρούνε, να βγούνε αυτά τα δύο μέρη από το τέλμα των διαπραγματεύσεων και να προχωρήσουν σε μια άλλη διαδικασία που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Κάτι ακόμα για τη Λιβύη προσθέτω. Έχουν γίνει εγκλήματα ε, φρικτά και συνεχίζουν να γίνονται εγκλήματα. Τόσο από τις πλευρές που μετέχουν στον ε, εμφύλιο πόλεμο, αλλά και όσον αφορά το εμπόριο ανθρώπων, τη διακίνηση ανθρώπων. Και εδώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ευθύνες πρέπει να κληθούν οι υπεύθυνοι να δώσουν εξηγήσεις για τις ενεργειές τους. Τι κάνετε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο. Και όσον αφορά τις μεγάλες ε, παγκόσμιες δυνάμεις, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το δικαστήριο μέχρι ότου να έχει και τη στήριξη των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας, θα έχει δυσκολίες επιχειρησιακές σημαντικές στην άσκηση του έργου του. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν ποια βήματα έχουν γίνει ως προς αυτό, κυρίως απέναντι στις ΗΠΑ, και ακόμη μια φορά να σας πω ότι σας στηρίζουμε απόλυτα. Να μην ακούτε αυτούς που λένε πρέπει να ελαφριθεί η πίεση προς την Αφρική γιατί σε άλλα μέρη δεν έχουν γίνει αρκετά. Όχι, να μην μειώσετε την πίεση, να μην υποχωρήσετε στις διπλωματικούς εκβιασμούς που προέρχονται από αλλού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Κριστόλτο. Πριν δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της υπηρεσίας της εξωτερικής δράσης, ήθελα και εγώ να διατυπώσω κάποιες ερωτήσεις προς την κυρία Βενσούντα. Ξεκινώ λέγοντα ότι για μα ο καλύτερο τρόπο να εξυπηρετηθούν ανθρώπινα δικαιώματα από την προοπτική του διεθνού δικαίου είναι αυστηρά η διατήρηση της ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητα η αποφυγή κάθε κατάχρησης και παρέλκυσης της αποστολής του Διεθνούς Δικαστηρίου. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι όσοι είμαστε μέλη της Επιτροπής μας. Ιδιαίτερα για την υπηρεσία εξωτερική δράση θα το αναφέρω αυτό, αλλά θα ήθελα και επί τη ευκαιρία να πω, μια και είναι εδώ η κυρία Μπενσουντά, να τυπώσω τι εξή ερωτήσεις. Πρώτον, πολύ διατυπώνων ε, επικρίσεις στο καταστατικό της Ρώμης, σε σχέση με την περιγραφή των εγκλημάτων, ότι δεν είναι Δεν υπήρξε από ό,τι φαίνεται συνένεση μεταξύ κρατών, όμως τώρα μπορεί αυτό να ισχύει, μπορεί να υπάρχει συνένεση, εσείς τη λέτε. Και για τη Γάζα και την Παλαιστίνη και τη διαδικασία για τις ένταξεις της ως συμβαλόμενο μέρος ε, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επικρίσεις διατυπώθηκαν και από το Ισραήλ. Δεδομένου ότι επικαλούμενο το 2013 η Παλαιστίνη τον Ιανουάριο του 2015 ξεκίνησε τη διαδικασία και καταήγγειλε παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Αλλά τρεις μήνες νωρίτερα είχε αναβαθμιστεί από τη Γενική Συνέλευση το καθεστώς της Παλαιστίνης σε μη μέλος κράτος παρατηρητή. Και χαρακτηρίστηκε αυτή η αναγνώριση ως, έχουσα, ως μη έχουσα αναδρομική ιστή. Η Παλαιστίνη λοιπόν από εκεί και πέρα μπορεί να ε, ενταχθεί στο καταστατικό της Ρώμης. Αυτές είναι οι επικρίσεις που έχουν απευθυνθεί. Ε, θα ήθελα να δώσετε απαντήσεις. Γιατί μπορεί να αποτελέσει η αναδρομική αυτή ε, αναγνώριση ευκαιρία για ηγέτες των Παλαιστινίων να προωθήσουν πολιτικά, πολιτικές επιδιώξεις. Τώρα θα παρακαλώ τον κύριο Κρίστιαν Μπέρμαν από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβει το λόγο και στη συνέχεια κυρία Μπενσοντά για να απαντήσει παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, επαναλαμβάνουμε από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ότι υπάρχει αυτή ε, το ότι το γεγονός ότι, ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση και η συνεδρίαση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς δεν μπορούμε παρά να υπογραμμίσουμε την ε, σαφή υποστήριξη στην, ε, στο Εθνικό Δικαστηρίο και την, τον αγώνα για την καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Το ΔΟΠΟΔΟ είναι ένα πολύ σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο για την καταπολέμηση της ατιμορρησίας και την επιβολή ενός διεθνούς, ε, μιας διεθνούς στο δίκαιο για αυτό το, το λόγο είναι πολύ σημαντικό σε εταίρο για μα το δοπουδό, για την Ευρώπη εν γέννη. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εξαίρετες ε, σχέσεις συνεργασίας ε, με την υπηρεσία μας. Το δικό σας το γραφείο, το γραφείο του Λέτου Εισαγγελέα, συνεργάζεται πολύ καλά με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και βεβαίως ε, αξιοποιούμε τις δυνατότητες συνεργασίας που μας προσφέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να διατυπώσει ερώτηση. Όχι. Κύριε Μπενσουντά, έχετε το λόγο. Και θα ήθελα να πείτε και δύο λόγια για την στρατιωτική δράση στη Συρία. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσει σας. Κάμποσε, Αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. Πρώτη ερώτηση. Για την Ουκρανία. Ποια είναι η κατάσταση. Όπως είπα και στην παρουσίασή μου, έγινε δεύτερη δήλωση βάσει της οποίας η Ουκρανία δέχτηκε τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Στην πρώτη δήλωση ε, καλύπτονταν τα γεγονότα της Μεϊντάν. Επρόκειτο για ένα προσωρινό στόχο με τη δήλωση αυτή ήταν από Νοέμβριο του 2013 μέχρι το Φεβρουάριο του 2014. Κάλυπτε αυτά τα γεγονότα δηλαδή και μπορούσαμε μόνο να ασχοληθούμε με αυτήν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πρέπει να περιοριστούμε. Και δεν ήταν εύκολο για το δικαστήριο. Πολλά θέματα βέβαια τότε θέταμε γιατί να περιοριστούμε σε αυτό το χρόνο, αλλά πάντως η δήλωση μας περιόριζε χρονικά. Με την ε, δεύτερη όμως δήλωση που πήραμε τον προηγούμενο μήνα, ή αυτό το μήνα. Τι έγινε. Δέχεται την δικαιοδοσία πάλι από το Φεβρουάριο του 2014 και μετά, χωρίς λήξη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει επέκταση της προκαταρτικής εξέτασης και συμπεριλαμβάνει και άλλα γεγονότα, ακόμα και στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Άρα δηλαδή είναι ευρύτερη η δικαιοδοσία την ανακοίνωση τη σχετική την έκανα χτες που είπα ότι επεκτείνουμε την προκαταρτική εξέταση προκειμένου να καλύψουμε και άλλα γεγονότα. Θέλω επίσης να είμαι σαφής για τις προκαταρτικές εξετάσεις και να σας πω ότι δεν πρόκειται για έρευνα. Πρόκειται για συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά τα εγκλήματα και πρόκειται για ανάλυση των πληροφοριών αυτών. Αναλύουμε δηλαδή. Απαιτείται αξιόπιστη πληροφορία, όλες τις πληροφορίες τις διασταυρώνουμε και καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα. Κατά πόσο έχουν γίνει εγκλήματα, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, κατά πόσο υπάρχουν εθνικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην προκαταδική εξέταση, το κοιτάμε αυτό. Κοιτάμε επίσης και τη σοβαρότητα των αδικημάτων και μετά βλέπουμε κατά πόσο θα ήταν κατά της δικαιοσύνης αν παρεμβαίναμε σε βάρος της δικαιοσύνης. Μόνο μετά από τη διαδικασία αυτή αποφασίζουμε για τη συνέχεια, ανάλογα δηλαδή με τις πληροφορίες που έχουμε και την απόφασή μας την παίρνουμε μετά για να αρχίσουμε ή να μην αρχίσουμε την δικαστική έρευνα. Εκεί βρισκόμαστε με την Ουκρανία τώρα. Όσον αφορά την Παλαιστίνη τώρα, το αναφέρατε και αυτό και πρόκειται για την ίδια διαδικασία. Στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε, δηλαδή συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες, τις αναλύουμε και μετά θα αποφασίσουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλες τις προκαταρτικές εξετάσεις και κυρίως για την κατάσταση στην Παλαιστίνη να εξαντλήσουμε τις πληροφορίες που έχουμε και να τις αναλύσουμε όλες πριν καταλήξουμε σε απόφαση για να αρχίσουμε να μην αρχίσουμε δικαστική έρευνα. Και στην υπηρεσία μου το είπα από την αρχή ότι έχω καλέσει όλες τις πλευρές να στείλουν ό,τι πληροφορίες έχουν. Όπως είπα και στην αρχή, στην παρουσίασή μου, όλες οι πλευρές μπορούν να έρθουν και να δώσουν πληροφορίες και το κάνουν. Είναι καλό αυτό γιατί όπως πάλι είπα πριν, είναι πάντα προτιμότερο να έχουμε όσο γίνεται πιο πλήρη εικόνα και από κάθε δυνατή πηγή κατά τη διάρκεια της προκαταρτικής εξέτασης. Ήδη λοιπόν συμβαίνει αυτό. Με εργαζόμαστε. Είναι μια, θα έλεγα, χωρίς ε, φασαρία διαδικασία στο προσκήνιο, αλλά γίνεται επεξεργόμαστε τις πληροφορίες που έχουμε τώρα. Για επίσκεψη στην Παλαισίνη, ναι, ήδη έχουμε ζητήσει και από την Παλαιστινιακή Αρχή και από το Ισραήλ να επισκεφθούμε την περιοχή. Θα πάει μια αποστολή μας και πιστεύω ότι θα είναι θετικό. Μάλλον μέσα στους επόμενους μήνες θα γίνει ή αυτόν, δεν ξέρω. Πρέπει να μας απαντήσουν πρώτα. Κάτι άλλο που θέλω να πω για την προκαταρκτική εξέταση είναι ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Εξαρτάται από τα γεγονότα και από τις συνθήκες. Πρόκειται για συγκέντρωση πληροφοριών, όπως σας είπα, ανάλυση των πληροφοριών. Δεν πρόκειται για έρευνα. Είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε χρονοδιάγραμμα, να πούμε δηλαδή ότι αρχίζω σήμερα και θα τελειώσω τότε. Εξαρτάται από το τι πληροφορίες θα μας έρθουν για να μπορέσουμε να τηρήσουμε και τα κριτήρια που έλεγα, να ξέρουμε αν υπάρχει διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο, αν ε, θα πληγεί η εθνική δικαιοσύνη στην περίπτωση που εμείς παρέμβουμε κτλ. Συρία τώρα. Όπως πολύ σωστά είπατε, δεν αποτελεί μέρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Δεν έχουμε δικαιοδοσία δηλαδή εκεί και δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην κατάσταση στη Συρία αυτή καθ' αυτή. Όμως γνωρίζουμε ότι όσον αφορά το ISIS, το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος και τα εγκλήματα τα οποία λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια της Συρίας και του Ιράκ, γνωρίζουμε ότι στις γραμμές του ISIS υπάρχουν και άτομα που προέρχονται από χώρες οι οποίες αποτελούν μέρο του Δουπουδού και δρούν και σε βάρος και πολιτών χωρών που συμμετέχουν στο ΔΟΠΟΔΟ. Συνεπώς, επί των ατόμων αυτών έχουμε δικαιοδοσία. Βέβαια εδώ πρέπει να κοιτάξουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε κατά πόσο οι χώρες αυτές, κάθε αυτές των οποίων οι εμπλέκονται στις εγκληματικές αυτές δραστηριότητες, κάνουν κάτι. Γιατί όπως ξέρετε, η δικιά μας η δικαιοδοσία δεν αντικαθιστά τη δικαιοδοσία χωρών μελών, τη συμπληρώνει. Εμείς κοιτάμε απλώς κατά πόσο είναι όντως σωστές οι διαδικασίες ή όχι. Άρα πρώτα πρέπει να δούμε αυτό, τι κάνουν δηλαδή χώρες οι οποίες είναι μέρος του δουπουδού. Δεύτερον, κοιτάμε την ιεραρχία. Στην ιεραρχία δηλαδή, τι θέση έχουν οι υπεύθυνοι. Ζητούμε λοιπόν πληροφορίες για να μπορέσουμε να αναλύσουμε περισσότερο. Και ζητάμε τη βοήθεια των χωρών αυτών, των οποίων οι πίκοοι έχουν ενταχθεί στο έσις. Τότε βλέπουμε τι δυνατότητες έχουμε να διώξουμε και να δικάσουμε τους υπεύθυνους. Έρχομαι τώρα στη Νότια Αφρική, γιατί αναφερθήκατε σε αυτό και στην αποτυχία της Νότιας Αφρικής να συλλάβει τον πρόεδρο του Σουντάν. Μα πρόκειται για μια υποχρέωση ε, συμβατική που έχει η χώρα. Αν το δικαστήριό μας ε, διώκει κάποιον και βρεθεί στην επικράτεια μιας χώρας μέρους, το ότι η χώρα αυτή έχει την ευθύνη να συλλάβει τον ε, καταζητούμενο και να τον παραδώσει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κάτι που δεν έγινε στην περίπτωση Νότιας Αφρικής. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε ως υπηρεσία. Ενημερωθήκαμε για την αποτυχία αυτή της Νότιας ε, Αφρικής, ενώ τους είχαμε ενημερώσει και το εθνικό του σύστημα και ήξεραν ότι ο πρόσβαση έπρεπε να συλληφθεί και να παραδοθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τελικά, την ευθύνη την έχει το σώμα των χωρών μελών του ICC, <clears throat> αλλά και το Συμβούλιο Ασφαλείας. Για να δούνε πώς θα αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο ζήτημα όταν μία χώρα μέλος παραβιάζει τελικά τις οδηγίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει και το Συμβούλιο Ασφαλείας. Έρχομαι τώρα στις επόμενες ερωτήσεις σας. Με ρωτήσατε τη γνώμη μου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. που δεν κάνει δήλωση, ενώ συνήθως κάνει για την ε, επικύρωση της Παλαιστίνης, της Συμβαστής Ρώμης. Αλλά αυτό είναι πολιτικό θέμα και εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. θα έλεγα να ρωτήσετε ποιος είναι ο λόγος. Προτιμώ να μην σχολιάσω από αυτού. Για τις πολιτικές αποφάσεις δηλαδή. Άλλον διεθνών οργανισμό. Έπειτα ρωτήσατε πόσο καιρό θα πάρει. Σε αυτό απάντησα λίγο πολύ. Σας είπα ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει ημερομηνία λήξη στι προκαταρκτικές εξετάσει. Δεν μπορούμε να πούμε θα κρατήσει τόσο. Γιατί εξαρτάται από τα γεγονότα, από τι συνθήκε, από τη συλλογή πληροφοριών και την ανάλυση του. Για τη συνεργασία, επίση είπα ότι όλε οι πλευρέ αποφάσισαν να συνεργαστούν με την εισαγγελία. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε συναντήσεις και θα δούμε τελικά πόσο χρόνο θα πάρει. Και για την επίσκεψη σας είπα ότι προσπαθούμε να πάμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ρωτήσατε επίσης για τη διαδικασία. Υπάρχει η επικύρωση, αλλά Ακόμα και με δήλωση πρόκειται για τα εγκλήματα, τα δικήματα τα οποία έλαβαν χώρα το καλοκαίρι που μας πέρασε στην Γάζα, αλλά και πάλι είναι ευρύτερο με την έννοια ότι ζητάει από το δικαστήριο να επικεντρωθεί στα δικήματα αυτά, αλλά και στην επικράτεια της Παλαιστίνης, αλλά και σε πολίτες της Παλαιστίνης. Και αυτό είναι που μας επιτρέπει να κοιτάξουμε ευρύτερα όλα τα δικήματα τα οποία κάζεται ότι έλαβαν χώρα. Αυτό κάνουμε λοιπόν. Δεν περιοριζόμαστε μόνο στα γεγονότα του καλοκαιριού που πέρασε. Πριν, όχι του, πιο πριν ακόμα, το 14. Αν δεχόμαστε πίεση, όχι. Δεν δεχόμαστε πίεση. Αλλά ακόμα και αν υπήρχε πίεση, δεν πρόκειται να με επηρεάσει. Εγώ κάνω τη δουλειά μου. Αυτό κάνω. Συρία. Εξήγησα νομίζω για τη Συρία, σας είπα και για το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος και για την δικαιοδοσία που μπορούμε να έχουμε επί υπηκών των χωρών μελών μας. Όσον αφορά τώρα... Τώρα για την παραπομπή στο διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο μας το ζητάνε. Δεν πάμε εμείς στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να πούμε θέλουμε. Και ακόμα αν μας έρθει κάποιο τέτοιο αίτημα, εμείς δεν το κάνουμε αυτόματα, το αξιολογούμε πρώτα. και προετοιμαζόμαστε. Το κάναμε για τον Ταφούρ στο Σουδάν, το κάναμε για τη Λιβύη πριν αναλάβουμε την υπόθεση. Αλλά οι δυνατότητες τις οποίες αναφέρεστε είναι το κατά πόσο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παίρνει την πρωτοβουλία για τη Συρία. Όχι. Ή που θα υπάρξει αίτημα από το Διεθνές Δικαστήριο, θα υπάρχει δήλωση αναγνώρισης της δικαιοδοσίας. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Για το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Και εσείς αναφερθήκατε στην Παλαιστίνη, απάντησα νομίζω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάντως που με ενθαρρύνετε. Να μην παρετούμε. Μα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν μου περνάει από το μυαλό. Αναφερθήκατε και στο θέμα της τρομοκρατίας. Και γιατί δεν ορίζεται συγκεκριμένα στο κείμενο της Ρώμης. Οι πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση της τρομοκρατίας είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας βάση του κειμένου της Ρώμης. Αν υπάρχει λοιπόν επίθεση, δεν αναφέρεται ε, ρητά ως τρομοκρατική πράξη, αλλά δεν σημαίνει ότι το δικαστήριο δεν μπορεί να εξετάσει τέτοια εγκλήματα εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις. Γιατί εμπίπτουν σε άλλες κατηγορίες, για παράδειγμα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δολοφονίες, καταστροφές ή άλλο είδους εγκλήματα. Δεν εμποδίζει δηλαδή αυτό το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να δράσει και σε περιπτώσεις τρομοκρατίας, εφόσον έχει δικαιοδοσία. Αναφερθήκατε στη δήλωση επίσης που ενθαρρύνω λίγο πολύ την ε, Παλαιστίνη. Οι επικρίσεις είναι άδικες και ασφαλμένες. Δεν υπήρξε ενθάρρυνση από τη δικιά μου την πλευρά. Όταν στα τέλη του 2013 η Παλαιστίνη πήρε το καθεστώς από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Πολλοί είπαν ότι τώρα που άλλαξε το καθεστώς της Παλαιστίνης στον Οιέ, τότε και εγώ θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω τη δήλωση του 2009 και να αναλάβω την Παλαιστίνη. Έγιναν ένα σωρό συζητήσεις ότι αυτόματα το γραφείο μου θα έπρεπε να αναλάβει την υπόθεση αυτή δεδομένη της δήλωσης που είχε γίνει το 2009. Και γι' αυτό και θεώρησα ότι θα έπρεπε να υπάρξει σαφήνεια. Να βγω δηλαδή και να πω ότι δεν λειτουργεί αναδρομικά το πράγμα, επειδή έγινε το 2009. Αυτά γίνανε το 2012 και όταν έγινε η δήλωση, τότε δηλαδή, το 9, δεν είχε το καθεστώς ε, που απέκτησε μετά η Παλαιστίνη στα Ηνωμένα Έθνη. Τίποτα άλλο δεν είπαμε. Πάντα λέγαμε ότι επρόκειτο για το καθεστώς της Παλαιστίνης στον ΟΙΕ. Τίποτα άλλο. Και αυτό προσπαθήσαμε να πούμε ότι το καθεστώς που είχαν το 2009 στον ΟΙΕ άλλαξε. Αυτό είπαμε. Τώρα βρίσκεται σε μια διαφορετική κατηγορία η Παλαιστίνη, βάσει της οποίας μπορεί να επικυρώσει τη Ρώμη όπως και οποιαδήποτε άλλη. Οποιοδήποτε άλλο σχετικό κείμενο. Ήμασταν σαφείς. Είπαμε ότι έχει να κάνει με το καθεστώς που έχει η Παλαιστίνη στον ΟΗΕ. Τίποτα άλλο. Και σημειώσαμε ότι άλλαξε αυτό με την ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του το 2012. Και ήταν ανάγκη νομίζω το γραφείο μου να κάνει αυτή την αποσαφήνιση. Δεν πρόκειται για ενθάρρυνση από τη δικιά μας την πλευρά. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Δεν ενθαρρύνουμε κανέναν. Φυσικά η οικουμενικότητα είναι πολύ σημαντικό για τη Ρώμη. Γιατί τότε θα αποφύγουμε όλες αυτές τις κατηγορίες για δίπλες προδιαγραφές, για ένα μίξει κτλ. Η οικουμενικότητα είναι καλό. Και ως αξιωματούχος θα έλεγα οποιοδήποτε μέρος δεν συμμετέχει να συμμετάσχει. Στη συγκεκριμένη πάντως περίπτωση της Παλαιστίνης δεν χρειάστηκε εγώ να ενθαρρύνω κανέναν, δεν το έκανα, αλλά ήταν σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε μετά τις κατηγορίες που έλεγαν ότι το γραφείο μας ε, ή εγώ αποφεύγουμε να αναλάβουμε την Παλαιστίνη, αφού είχε αλλάξει το καθεστώς και έπρεπε να το πω. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σπουδαία η ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα που έχετε σε εκκρεμότητα και βεβαίως μην διστάσετε ποτέ αν θεωρήσετε ότι μπορούμε να σας στηρίξουμε. ελπίζουμε ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα και σε σχέση με το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή. Σε ευχαριστούμε και πολύ καλή επιτυχία στη δουλειά σας.